Συνεχίζεται η συνεδρίαση. Τα χθεσινά πρακτικά έχουν διανεμηθεί ήδη. Δεν ξέρω αν υπάρχουν παρατηρήσεις. Πρέγω. Νο. Α, νο. Un'abitudine alzare il catch the eye. In questo caso... Ah, λοιπόν.